So, dear colleagues, um, are we begin just slightly late on this. Ξεκινούμε, αγαπητοί συνάδελφοι, με μια μικρή καθυστέρηση στο 23, καταρχάς, στο σημείο 23. Καλώς ήρθατε τους συναδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και Δικαιοσύνης. Καλώς ήρθατε, κύριε Σόφερ. Πρώτη φορά, αν δεν απατώμε, στην Επιτροπή μας και τους άλλους δύο βέβαια συναδέλφους της Γενικής Διεθνής Εσωτερικών. Ας ξαναρχίσουμε λοιπόν. Καλό είναι να να συστηνόμαστε πριν ξεκινήσουμε. Έχουμε διάφορα θέματα. Σήμερα είχαμε τον Υπουργό της Μετανάστευσης της Ελλάδας και άλλους την προηγούμενη εβδομάδα. Πολλά θέματα λοιπόν που συζητούμε για την πολιτική ασύλου το Συμβούλιο, οι βουλευτές ενδιαφέρονται ιδιαίτερως. Στο συγγνώμη που δεν έχουμε πολλούς ε, συναδέλφους ε, παρόντες, γιατί με το τέλος και τη θητείας έχουν διάφορες υποχρεώσεις. Μεταρρύθμιση του Δουβλίνου, λοιπόν, είναι το θέμα μας. Ήμουν και στο τελευταίο άτυπο συμβούλιο δικαιοσύνη και εσωτερικών και τέθη το ζήτημα ότι κάνουμε τα προσωρινά μέτρα. Μέχρι ότου να υπάρξει μια πλήρης μεταρρύθμιση, διαρθρωτική μεταρρύθμιση ή αν υπάρχουν προτάσεις ε, να αποσπάσουμε κάποια συγκεκριμένα κομμάτια από το σύνολο των μέτρων ή αν πρέπει η μεταρρύθμιση του Δουβλίνου να προχωρήσει μαζί με όλα τα άλλα συναφή ζητήματα. Αν και θα χρειαστεί ευελιξία σε σχέση με, τα άλλα, με τις άλλες προτάσεις. νόμι μετανάστευση, όλα αυτά τα ζητήματα. Το Δεκέμβριο λοιπόν ανακοίνωση για τη διαχείριση της μετανάστευσης και όλων των πτυχών της. Οδήγησε σε πολλές συζητήσεις που συνεχίζονται. Επιτροπή, Προεδρία. Ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο έχει προχωρήσει ήδη, έχει αναθέσει σε διαφορούς συγκητές η Επιτροπή μας, όπως γνωρίζετε, να καταρτήσουν τα σχετικά έγγραφα. Άρα η θέση του Κοινοβουλίου είναι σαφής. Θέλουμε να μην διασπαστεί η ενότητα του αρχικού ή του κυρίου τουλάχιστον κορμού των μέτρων. Από την άλλη θέλουμε να γίνει και μια ουσιαστική συζήτηση. Ε, ενισχυμένη συνεργασία λέμε. Το θέμα της ειδική ε, πλειοψηφία βέβαια μας απασχολεί εφόσον δεν ε, περάσει, ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο γενικά. Είμαστε πεπισμένοι όμως και αποφασισμένοι να προχωρήσει ε, ενιαίο το πακέτο. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τη δική σας παρουσίαση για τις προσωρινές ρυθμίσεις. ή αν υπάρχουν κάποιες προσωρινές διευθυντήσει. Ο Μιχαήλ Σότερ, λοιπόν, από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Εσωτερικών και ο κύριος Περλανκού επίση από την Προεδρία, από τη Ρουμανική Προεδρία βέβαια. Αλλά καλώς ορίζω πρώτα τον Μιχαήλ Σότερ. Παρακαλώ, να έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή σας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να συζητήσω μαζί σας το θέμα αυτό, το οποίο είναι σημαντικό και από ό,τι καταλαβαίνω ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους ευρωβουλευτές. Όπως είπατε, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα άτυπο συμβούλιο στο Βουκουρέστι. Μάλιστα ήσασταν παρόν στην ε, συζήτηση αυτή ε, που είχε να κάνει και με τις προσωρινές ρυθμίσεις. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις εμπειρίες του καλοκαιριού. Ο πρόεδρος Γιούνκερ αναφέρθηκε σε αυτές ε, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης. Αναφέρθηκε σε αυτές και είπε ότι δεν έχουμε ε, το περιθώριο να βρίσκουμε λύσεις ad hoc ε, με την άφηξη κάθε νέου πλοίου. Όσον αφορά τις δικές σας παρατηρήσεις, ανέφερε επίσης ότι χρειαζόμαστε μια μακροπρόθεσμη λύση και μόνιμη αλληλεγγύη. Απότερος στόχος, ο σαφής στόχος, είναι να έχουμε τέτοιες μόνιμες λύσεις. Στο μεταξύ όμως θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε την παρούσα κατάσταση. Και ενώ συνεχίζουμε τη συζήτηση σχετικά με το πώς θα προχωρήσουμε με τον κανονισμό του Δουβλίνου, συζητάμε και την ανάγκη προσωρινών ρυθμίσεων. Και όπως είπατε, είναι κάτι που αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής του Δεκεμβρίου για τη μετανάστευση. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται ότι στόχος είναι όχι να αντικαταστήσουμε, να υποκαταστήσουμε τις εργασίες ε, για τη μεταρρύθμιση του Δουβλίνου, ούτε να αναβάλουμε την πρόοδο Στόχο έχουν οι ρυθμίσεις αυτές να αποτελέσουν γέφυρα μέχρι να έχουμε τις μόνιμες ρυθμίσεις. Και γι' αυτό επισημάνθηκε ότι η δουλειά πάνω στις προσωρινές ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε όλους να συμμετάσχουν. Οι προσωρινές αυτές ρυθμίσεις θα σημάνουν ότι ήδη τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να ε, επιδείξει αλληλεγγύη στα κράτη-μέλη που το ζητούν. Θα πρέπει να φροντίσουμε αυτό να γίνει με τρόπο που να διασφαλίζει και την πρόληψη δευτερογενών κινήσεων. Είδαμε ε, με τις αφήξεις στη Μεσόγειο ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει εάν αποφύγουμε μία μη συντονισμένη προσέγγιση. Εάν δημιουργήσουμε ένα ε, κοινά συμπεφωνημένο εθελοντικό πλαίσιο. Αντί λοιπόν για λύσεις ad hoc, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια οργανωμένη μορφή συντονισμού. Οι πρόσφατες εμπειρίες μας από το Sea-Watch 3, το πλοίο, ήταν ε, ένα θετικό βήμα. Είχαμε μία δοκιμή, αν το θέλετε, της προσέγγισης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είχαμε δηλαδή καταγραφή και μετεγκατάσταση των ε, ανθρώπων και οι περισσότεροι από τα, τους 42 ανθρώπους που αποβιβάστηκαν από το Sea-Watch 3 αυτή τη στιγμή μεταφέρονται σε άλλα κράτη-μέλη. Αυτό πώς θα λειτουργήσει πιο γενικά. Εάν βρίσκεται υποπίεση ένα κράτος μέλος ή όταν είναι απαραίτητο να υπάρξει συμβολή στην γρήγορη αποβίβαση μετά από μια διάσωση, ένα κράτος μέλος μπορεί να αναζητήσει βοήθεια από άλλα κράτη-μέλη ε, που να περιλαμβάνει την μεταγκατάσταση. Επίσης μπορεί να διασφαλιστεί η συνδρομή της Επιτροπής και των σχετικών οργανισμών σε απάντηση τέτοιου αιτήματο, όπως είδαμε στα πιο πρόσφατα παραδείγματα, τα κράτη-μέλη θα αναφέρουν το συγκεκριμένο είδος ε, στήριξης που μπορούν να παράσχουν με προηγούμενο προγραμματισμό και με μέτρα αλληλεγγύης. Τα μέτρα αλληλεγγύης που προσφέρουν τα κράτη-μέλη αυτά θα πρέπει να συνδυάζονται με τις δράσεις του κράτους μέλους που είναι εκτεθειμένο στη συγκεκριμένη κατάσταση, το κράτος μέλος που βρίσκεται υποπίεση και αναζητάει βοήθεια. Το κράτος μέλος όπου αποβιβάζονται τα ε, άτομα αυτά. Λαμβάνει λοιπόν μέτρα και θα πρέπει να βρούμε μια σωστή δομή συντονισμού για να ανταποκριθούμε στα αιτήματα κρατών μελών. Αυτές είναι οι εμπειρίες μας από τους τελευταίους μήνες. που μπορεί να φανούν χρήσιμες τελικά. Μαζί με τους οργανισμούς θέλουμε να δημιουργήσουμε ε, πίνακες για απλοποίηση και συντονισμό της βοήθειας. Επίσης, είναι χρήσιμο να πραγματοποιείται συντονισμός όχι μόνο εδώ, αλλά και επιτόπου. Το πρόσφατο παράδειγμα του Sea-Watch ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οργανισμοί είχαν ανθρώπους επιτόπου που συνεργάζονταν με τα κράτη-μέλη που είχαν ανταποκριθεί στο αίτημα του κράτους μέλους υποπίεση. Ήταν λοιπόν πολύ χρήσιμη αυτή η εμπειρία. Τέλος, είναι πολύ σαφές ότι θα πρέπει να υπάρχει χρηματοδοτική υποστήριξη από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διευκολυνθεί όλη η διαδικασία. Η οικονομική στήριξη λοιπόν θα πρέπει να παρασχεθεί και θα παρασχεθεί στα κράτη-μέλη που θα προσφερθούν να συνδράμουν στην μετεγκατάσταση με τον τρόπο αυτόν. Ήδη έχει διατεθεί τέτοια οικονομική βοήθεια μέσω του ε, Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης. Στις πρόσφατες συζητήσεις ε, στην Κορεπέρ και στο άτυπο Συμβούλιο, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι είναι διατεθειμένη να συνεχίσει να υποστηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου αυτού, λαμβάνοντας υπόψη και τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό είναι χρήσιμο που βρίσκομαι εδώ σήμερα για ε, τούτη την ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ενδιαφέρον του και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι οι δράσεις μας πάνω στι προσωρινές ρυθμίσεις δεν θα πρέπει να υποκαταστήσουν ένα σταθερό και σύγχρονο νομοθετικό ε, πλαίσιο ε, με βάση τα συμπεράσματα που έχουμε βγάλει τα τελευταία χρόνια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σότερ. Πριν περάσουμε στη συζήτηση και τις ενδεχόμενες ερωτήσεις, ε, θα ήθελα να ακούσουμε τη Ρουμανική Προεδρία. Είπατε αν κατάλαβα καλά, ότι ακολουθεί διαφορετική γραμμή η Ρουμανική Προεδρία σε σχέση με την Αυστριακή Προεδρία. Θα το δούμε και απευθείας βέβαια, αλλά θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας απόψεις. Παρακαλώ. Thank you very Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Από την αρχή θέλω να σας πω ότι η αρχή που μας καθοδηγεί είναι να είμαστε ένα έντιμο διαμεσολαβητή. Είμαστε πεπισμένοι ότι οι λύσει ad hoc το μόνο που μπορούν να προσφέρουν είναι μία απάντηση σε μία δεδομένη κατάσταση. Άπαξ, τα νούμερα ε, μειώνονται σημαντικά. Εξακολουθούν όμω να υπάρχουν μεταναστευτικέ ροέ προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές φορές ε, ε, μιλάμε για πολύ επικίνδυνα ταξίδια στη Μεσόγειο που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Είναι και παραμένει πρόκληση το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να την αντιμετωπίσουμε προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται σίγουρα όμως μια κοινή αντίδραση και πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι αλλά και να γνωρίζουμε πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους καταστάσεις με δομημένο τρόπο, αποδεικνύοντας ότι είμαστε σε θέση να αντιδρούμε με αλληλεγγύη. Έτοιμος δημοσιολαβητής ε, σημαίνει ότι η Προεδρία άκουσε την έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση της Κορεπέρα αρχές Ιανουαρίου για να βρεθεί μια λύση στην πρόσφατη κατάσταση στη Μάλτα, όπου είχαμε μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με αποτέλεσμα 49 μετανάστες να αποβιβαστούν εκεί. Οκτώ κράτη-μέλη πρότειναν ε, να πάρουν το άσυλο από τη Μάλτα. Πέντε αιτήσει ήταν δεκτέ η Μάλτα, η, συγγνώμη, η Ρουμανία συγκεκριμένα. Και αυτό δείχνει και αλληλεγγύη αλλά και υπευθυνότητα. Όταν το Sea Watch 3, δεύτερο σκάφος, ε, αποβίβασε κάποια άτομα στην Ιταλία, έξι κράτη-μέλη προσφέρθηκαν να πάρουν τον δεσάσιλο από την Ιταλία και πάλι η Ρουμανία ήταν μεταξύ αυτών δέχθηκε να φιλοξενήσει μια οικογένεια πενταμελή εξαμελή. Και όλα αυτά αποδεικνύουν ότι ορισμένα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ρουμανία, αντιλαμβάνονται την ανάγκη για αλληλεγγύη και την ανάληψη ευθύνης όταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει μια ειδική κατάσταση. Ταυτόχρονα σε μια προσπάθεια αντικατάσταση αυτών των ad hoc από μια πιο συντονισμένη προσέγγιση, λάβαμε υπόψη την έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την ανάπτυξη προσωρινών ρυθμίσεων για πραγματική αλληλεγγύη και υπευθυνότητα με την επιφύλαξη της συζητήσης ε, ως για τον κανονισμό του Δουβλίνου. Θα πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουν διεξαχθεί αρκετές συζητήσεις και το ζήτημα συζητήθηκε ανεπίσημα σε επίπεδο κορεπέρ και άτυπου υπουργική διάσκεψη ε, των Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνη ε, στι 7 του μήνα στο Βουκουρέστι και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Στόχος μας είναι να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα θα αποδείξει αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να ανταποκριθεί με καλύτερο τρόπο στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ανθρώπων από τη Μεσόγειο. Τις επόμενες εβδομάδες αποσκοπούμε στη συνέχιση των συζητήσεων σε επίπεδο πρέσβεων, κορεπέρ, με την πρόθεση να διερευνήσουμε και να συζητήσουμε διάφορα ζητήματα από τη στιγμή δηλαδή της καταχώρησης της αίτησης ε, παροχής ασύλου μετά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μέχρι την πιθανή ανακατανομή σε άλλα κράτη. Στα κράτη όμως τα οποία συμμετέχουν εθελοντικά σε αυτό το σύστημα. Και μια σημαντική πτυχή είναι και αυτή των, της επιστροφής στη χώρα καταγωγής για μετανάστες που δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας. Όλες οι πτυχές αυτές θα συζητηθούν ενδελεχώς με στόχο να βρεθούν επιχειρησιακές λύσεις και η Ένωση να έχει στη διάθεσή της ένα σύστημα που να τη επιτρέπει να αντιδρά με κοινό τρόπο και να ε, εγγυάται ξεκάθαρες διαδικασίες ε, διεκπαιρέωση αιτήσεων ασύλου και επιστροφών ενδεχομένω. Σε στρατηγικό επίπεδο θέλουμε να δούμε και στο Βουκουρέστι στην προσεχή συνεδρίαση της 24 Μαρτίου, όπου όλα τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο τους από την επιχειρησιακή σκοπιά περισσότερο, με στόχο να έχει εξευρεθεί το στόμα των δετών μια καλή λύση. Με βάση την έκβαση της συνεδρίας αυτής η Προεδρία θα συζητήσει το θέμα και στη συνέχεια στο αρμόδιο, στο αρμόδιο επίπεδο. Θέλω να σας πω ότι η Προεδρία αντιλαμβάνεται πλήρως τη σημασία Τη συζήτηση αυτής και του θέματο αυτού και δεσμευόμαστε να αναζητήσουμε λύσεις, συνεργασία με όλους τους άλλους ενδιαφερομένους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank um, Σας ευχαριστώ πολύ. Μας είπατε ότι 8 κράτη-μέλη είχαν μπλακεί στην επίδειξη ελληνικής. Ποια ήταν αυτά? Ναι, δεν έχω τα ονόματα τους. Ίσως η Επιτροπή τα γνωρίζει. Σε ποια περίπτωση αποβίβασες εκεί, Μάλτα, Ιταλία. Το CY3 ήταν η τελευταία επιχείρηση στην Ιταλία. Γαλλία, Γερμανία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ρουμανία. Ωραία. Ερωτήσεις, Χουάν Φερνάντο. Θα ήθελα απλώς να απευθύνω μια απευθείας ερώτηση στο Συμβούλιο που προσωπείται από τη Ρουμανική Προεδρία, αλλά μην το πάρετε προσωπικά σας παρακαλώ, γιατί πεθαίνουμε στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο σε όλη αυτή την εντολή, στα πέντε χρόνια της εντολής, δεν φάνηκε να ασχολείται με την αλληλεγγύη, να προκρίνει την αλληλεγγύη. και για τις Ισραήλ και για τους ε, άσυλο. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι περιορίζεται η αλληλεγγύη μόνο σε προσωρινές ρυθμίσεις, με το άρθρο 80, είναι πολύ πιο ευρία η εντολή. Και καλύπτει όλη τη διαδικασία λήψη αποφάσεων για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ευρωπαϊκό δίκαιο ασύλου δηλαδή, ευρωπαϊκό δίκαιο μετανάστευσης. Εν αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη που όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουμε δει να εκδηλώνεται. Δεν υπάρχει. Πρώτα ήταν οι μόνες του Ιταλίου και η Ελλάδα, τώρα η Ισπανία. Και βλέπουμε ένα πινκ-πονγκ να προσπαθεί ο ένας να πετάξει τον μπαλάκι στο γήπεδο του άλλου πάνω από το δίχτυ. Αλλά αλληλεγγύη δεν βλέπουμε. Προσωρινές ρυθμίσεις δεσμευτικές με πλήρη τήρηση των όρων της εντολής. Ευρωπαϊκή πολιτική, ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πρέπει να τηρούνται. Ευχαριστώ. Κανείς άλλος. Για να σταθώ σε αυτά που είπε ο Μιχαήλ. Μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι τα ευρύτερα θέματα για το άσυλο και τα λοιπά, αλλά όλο αυτό το θέμα των προσωρινών μέτρων και το κενό Γιατί ακούμε, μαθαίνουμε ότι υπάρχουν προβλήματα και αδιέξοδα στη λήψη αποφάσεων. Η Γερμανία, η Γαλλία και το καθεξής. Το θέμα είναι τώρα τι κατεύθυνση θα προκύψει. Εάν χρειαστεί δηλαδή να κατακαιρματιστεί το σύνολο σε διάφορα κομμάτια, τι είδου προσωρινά μέτρα θα προχωρήσουν το Συμβούλιο, σε τι είδου προσωρινά μέτρα θα προχωρήσει το Συμβούλιο. γιατί είναι πολλά τα πολιτικά ζητήματα. Μικρός ο αριθμός των ε, ανθρώπων που αφορούν τα μέτρα αυτά, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντικό γενικά για την Ευρώπη το πώς θα αντιμετωπιστούν. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα στοιχεία σε σχέση με τα προσωρινά μέτρα. Τι μπορείτε να πείτε στο Συμβούλιο σαν πρόταση, γιατί δεν νομίζω ότι είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα αυτή η λύση, χωρίς να κάνει μια σοβαρή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αποβιβάσεις και τα λοιπά θέματα επίσης, που δεν έχουν συζητηθεί Πώ έχουν προχωρήσει όλα αυτά. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο ξέρουμε δεν τα έχει συζητήσει. Η Επιτροπή τα έχει μελετήσει. Και το γενικότερο θέμα, Δουβλίνο, άσυλο, διαδικασίε ασύλου. Γιατί μας ανησυχεί το ότι ακούμε πως πρόκειται για να γίνει μικρότερα κομμάτια το πακέτο των μέτρων. Πώς θα γίνει αυτό. Θα γίνει ένα διατύπωση από ό,τι ακούμε. Και τότε ανεξαρτήτως της ε, επανεγκατάστασης και τα λοιπά, ε, της Eurodac, ε, της υπηρεσία μπορεί να υπάρξουν διάφορες λύσεις. Έστω, αλλά το κύριο θέμα είναι εάν θα επαναδιατυπωθεί η βασική νομοθεσία. Τώρα δεν ξέρω αν μπορείτε να μου δώσετε απαντήσει σε αυτή την ερώτηση που είναι ρητορική μάλλον, αλλά... Μπορούμε να περιμένουμε κάποια ουσιαστική λύση πριν τις ε, ευρωεκλογέ ή απλώς θα φιλορροήσουμε μέχρι εκεί και μετά θα τα αφήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω τις ερωτήσεις που θέλετε. Είναι θεμελιώδους σημασίας και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται μια σταθερή μακροπρόθεσμη λύση με βάση τα συμπεράσματα των τελευταίων ετών και τις εμπειρίες από την κρίση που ζήσαμε. Η δουλειά πάνω στις προσωρινές ρυθμίσεις είναι πρακτικής φύσης. Όπως ανέφερα, είναι αντίδραση, όπως είπατε, στην πολιτική πίεση, στην αντιμετώπιση ε, συγκεκριμένων πλοίων που ψάχνουν τόπο να αποβάσουν τους ε, ανθρώπους που έχουν διασώσει. Είναι λοιπόν ένας τρόπος ε, να αντιμετωπίσουμε την πίεση αυτή. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βρει λύσεις, ε, έχει εντείνει τις προσπάθειές της. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Κάθε τέτοια εμπειρία το καλοκαίρι βρήκε μία λύση ad hoc, μη ικανοποιητική όσον αφορά την προσπάθεια που απαιτήθηκε σε κάθε τέτοια περίπτωση. Αυτό λοιπόν δεν αποτελεί βιώσιμη λύση. Η συζήτηση τώρα για τις προσωρινές ρυθμίσεις αποτελεί αντίδραση σε αυτά τα γεγονότα. Όπως όμως λέει και το όνομα, πρόκειται για προσωρινές ρυθμίσεις που δεν μπορούν να υποκαταστήσουν ε, πιο μακροπρόθεσμες και μόνιμες λύσεις. Όποιο λοιπόν και αν είναι το αποτέλεσμα των εργασιών αυτών, θα πρέπει να αποφύγουμε την παγίδα της ε, ε, υποκατάστασης των νομοθετικών ρυθμίσεων, διότι μόνο έτσι μπορούμε να βρούμε μια σωστή λύση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να εντείνει τις προσπάθειές της, δεδομένου του πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις εργασίες στην ομοθετική πλευρά. Ό,τι και να κάνουμε, οι προσωρινέ ρυθμίσει ε, δεν ε, υποκαθιστούν την νομοθετική δουλειά. Αποτελούν απλά ε, μια γέφυρα για τους επόμενου μήνες. Ελπίζω αυτό να απαντάει στην ερώτησή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος παρακαλώ. Μία σημαντική ερώτηση. Μπορεί να με διαβεβαιώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι προσωρινές ρυθμίσεις πράγματι θα αποτελέσουν μία γέφυρα για τη μεταρρύθμιση του Δουβλίνου και πώς λειτουργούν αυτές οι προσωρινές ρυθμίσεις. Um, well, Νομίζω ότι η απάντηση είναι ότι πρόκειται για τρέχουσες εργασίες και γι' αυτό, κατά την εισαγωγή μου, αναφέρθηκα στις μέχρι τώρα εμπειρίες μας. Πρόκειται για συνεχιζόμενες εργασίες και στην πιο πρόσφατη αποβίβαση που είχαμε, το Sea-Watch 3, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετείχε στον επιτόπου συντονισμό στην Ιταλία κατόπιν πρόσκλησης και με την πλήρη συνεργασία των Ιταλικών αρχών ε, ενώ συνεργαζόμασταν ταυτόχρονα επιτόπου με τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσέφεραν τη βοήθειά τους. Επίσης είχαμε κράτη-μέλη που υποσχέθηκαν να βοηθήσουν ε, και έτσι συντονίσαμε τις εργασίες τους τόπου. Αυτές οι εμπειρίες μπορεί να είναι χρήσιμες ε, στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχεδίων. Το πλεονέκτημα που μπορεί να καθησυχάσει νομίζω όλες τις πλευρές είναι ότι σε προηγούμενες περιπτώσεις κάποια κράτη-μέλη ε, δεσμεύτηκαν να βοηθήσουν, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις χρειάστηκε αρκετός χρόνος μέχρι οι δεσμεύσει τους να μεταφερθούν σε πραγματική ηλική βοήθεια. Η επιτόπου συμμετοχή λοιπόν με συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο στόχο είχε την επιτάχυνση των εργασιών, κάτι που είναι προς όφελος όλων. Ελπίζω αυτό να απαντάει στην ερώτησή σας. Σας ευχαριστώ κύριε Φράνς να ρωτήσω και τους δυο σας. Στο Συμβούλιο άκουσα τα κράτη-μέλη να θέτουν το αιώνιο ερώτημα της αλληλεγγύης. Στα, στις προσωρινές ρυθμίσεις, λοιπόν, τίθεται αυτό το θέμα της αλληλεγγύης και στην περίπτωση του Sea-Watch είχαμε τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, που βρέθηκαν υπό πολλή πίεση. Μιλάμε για σχετικά περιορισμένο αριθμό ανθρώπων. Ε, περιπτώσεις όμως ε, τις οποίες ε, κάποιοι πολιτικοί θα εκμεταλλευτούν στη ρητορική τους. Έχετε κάποια αίσθηση, κάποια κρατημέλη αντιδρούν με πιο θετικό τρόπο από ό,τι άλλα. Τι ακριβώς γίνεται στο Συμβούλιο. Διότι εδώ οι συνάδελφοι ακούν διάφορα στοιχεία. Αλλά ακούμε κάποια θετικά στοιχεία από το Συμβούλιο, κάποια πιο αρνητικά. Έχετε μια αίσθηση λοιπόν. Μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες σχετικές. επιτρέπετε να απαντήσω στα ρουμανικά. Cred că președinția română a dovedit de la bun început că s-a implicat. Din prima... Η Ρουμανική Προεδρία από την πρώτη στιγμή έδειξε ότι στηρίζει την Κομισιόν. Έχουμε εμπλακεί σε όλες αυτές τις δραστηριότητες ε, και ήμασταν σε μόνιμη επαφή από την αρχή με την Κομισιόν και τους εκτελεστικούς οργανισμούς για να λύσουμε το πρόβλημα των αποβιβάσεων αυτών ε, στη Μάλτα και την Ιταλία. Επίσης, ε, είχαμε ηγετική στάση και λάβαμε και την πρωτοβουλία να φιλοξενήσουμε ορισμένα άτομα, καλώντας ταυτόχρονα να μιμηθούν το παράδειγμά μας και τα άλλα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο. Καταλάβαμε πολύ καλά την έκκληση της Κομισιόν για τις προσωρινές ρυθμίσεις το Δεκέμβριο. Συνεχίσαμε και συνεχίζουμε τις συζητήσεις αυτές στο επίπεδο Κορεπέρ και Άτυπου Συμβουλίου και Οσύνης Εσωτερικών Υποθέσεων. Οι πρώτες μας εντυπώσεις είναι θετικές. Τα κράτη-μέλη αντιλαμβάνονται την ανάγκη να υπάρχουν αυτές οι προσωρινές ρυθμίσεις για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, το πρόβλημα των αποβιβάσεων. Διότι οι αποβιβάσεις αυτές, πρώτα απ' όλα, είναι ανθρωπιστικό ζήτημα. Μιλάμε για απώλειες ανθρώπινων ζώων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να δώσει απάντηση στο πρόβλημα αυτό. Επομένως, οι πρώτες μας εντυπώσεις είναι θετικές, εξού και μας παρακινεί περαιτέρω τρόπος με τον οποίο διεξάγονται οι συζητήσεις. Θέλουμε να τις συνεχίσουμε και από κοινού με την Κομισιόν θέλουμε να καταλήξουμε σε κάποιο είδου συνένεση. Σε ό,τι θα αφορά την αλληλεγγύη, την οποία μίλησε ο ξετοιμός βουλευτής, θεωρώ πως πάντοτε υπήρχε αλληλεγγύη. Υπήρχε αλληλεγγύη ακόμη και το 2015-2016, στο απόγειο της κρίσης. Ίσως βέβαια όχι στο επίπεδο που όλοι θα επιθυμούσαμε. Αλληλεγγύη όμως υπήρχε έδωσε μια κοινή απάντηση, υπήρξε μια κοινή αντίδραση από την Κομισιόν και σε ό,τι αφορά την μετεκατάσταση. Η Ρουμανία ήταν ένα από τα κράτη-μέλη που είχε αρχικά καταψηφίσει τις μετακαταστάσεις, αλλά ήταν το πρώτο κράτος μέλος που αποφάσισε να πάρει άτομα από την Ελλάδα. Ήταν το πρώτο κράτος μέλος ε, που έστειλε πυρογνώμονες στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, στα hot spot στην Ελλάδα και αλλού, για να βοηθήσει με την κατάσταση εκεί και ταυτόχρονα πιστεύουμε πως εξακολουθεί να γίνει ακόμη πολλή δουλειά για να υπάρξει αλληλεγγύη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρούμε ότι το πρόβλημα αυτό θα λυθεί, πρέπει να λυθεί, ιδίως σε νομοθετικό επίπεδο. Το είπε και ο Μάικλ άλλωστε πολύ σωστά. Εσείς όμως, θέλετε να ακολουθήσετε αυτή την προσέγγιση, να δοθεί το όλο θέμα ως πακέτο. Ε, αυτή είναι η δική σας πλευρά. Έχουμε και το Συμβούλιο που και αυτό έχει τη δική του ξεκάθαρη άποψη. Ε, εκεί ξεκινήσαμε από την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου να συζητάμε θέμα, ε, κάθε θέμα ξεχωριστά, διαδικασία παροχής ασύλου. Προσπαθήσαμε να βρούμε λύσεις ακόμη και στο ύψιστο επίπεδο, πολιτικό επίπεδο, επίπεδο Κορεπέρ. Και κάποιοι φάκελοι συστήθηκαν δύο φορές στην Κορεπέρ για να βρεθεί λύση. Θα μπορούσαμε λοιπόν να σημειώσουμε πρόοδο σε καθέναν από τους φακέλους, αν γνωρίζουμε ότι στο τέλος ε, θα ε, γίνουν δεκτά όλα αυτά ως πακέτο. Νομίζω πρέπει να αναγνωρίσει τι προσπάθειε που καταβάλει το Συμβούλιο από την αρχή και σίγουρα πρέπει να σημειωθεί πρόοδο σε κάθε μεμονωμένο φάκελο και βέβαια έχοντα κατά νου ότι στο τέλο θα τα δούμε όλα αυτά ω πακέτο. Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για τι διαδικασίε ασύλου, τα πράγματα προχωρούν καλά και πιστεύουμε ότι ζητήματα που αφορούν λεπτά θέματα όπως είναι η διαδικασία στα σύνορα και η τελική απόφαση, εκεί νομίζω ότι θα έχουμε πρόοδο. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κανονισμό του Δουβλίνου, είμαστε ακόμη στη φάση προβληματισμού σε επίπεδο Ρουμανική Προεδρία για να δούμε προ ποια κατεύθυνση θα πάμε. Γνωρίζετε ότι τον Ιούνιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μα έδωσε καθοδήγηση και ζήτησε να υπάρξει ισορροπία μεταξύ υπευθυνότητα και αλληλεγγύη. Και ξέρετε ότι αρκετέ Προεδρίε πριν από εμά κατέβαλαν τεράστιε προσπάθειες ε, για εξέβρεση ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο πτυχών, κάτι το οποίο επιδείχθη δύσκολο. Και αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πολιτική πραγματικότητα την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τώρα λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε ότι η νομοθεσία που προσπαθούμε να καταρτήσουμε δεν είναι για τώρα αλλά για το μέλλον. Επομένως πρέπει να είναι ποιοτική και ταυτόχρονα πρέπει να ανταποκρίνεται και στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Ελπίζω να απάντησα με επιτυχία στα ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίω ε, δεν αμφισβητήθηκε η πρόοδο, αλλά υπήρχε και στην Βουλγαρική Προεδρία αντίστοιχη ε, προόδο. και δυστυχώς, δυστυχώς είδαμε μια οπισθοδρόμηση κατά τη διάρκεια τη Αυστριακή Προεδρία. Τώρα με τη Ρουμανία βλέπουμε μια πιο θετική προσέγγιση. Με βεβαίω ότι όλοι μα θέλουν να δουν να συνεχίζεται. Είναι πολλά τα θέματα όμως και προκύπτουν πράγματα τα οποία δεν έχουμε συζητήσει επαρκώς. Προσωρινά μέτρα, α, γενικά τα θέματα του ασύλου. Ενώ εμείς στο Κοινοβούλιο τα συζητούμε διαρκώς. Μας βοηθάτε λοιπόν με την παρουσία σας εδώ και τις εξειδικευμένες γνώσεις. Σας ευχαριστούμε κύριε Σότερ. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Δικαιοσύνης, κύριε Μπελάτσου, εσάς και τις ομάδες σας βέβαια για το χρόνο που μας αφιερώσατε απόψε. And if the commissioner would like to come to the front, please. Και θα παρακαλέσω τον κύριο Επίτροπο να έρθει. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Η ώρα είναι πέντε. Έχουμε όμως ένα πολύ ωραίο θέμα, έτσι για να ολοκληρώσουμε την απόψηνή μας συνεδρίαση. Έχουμε και ένα, ε, μια μικρή δεξίωση μετά για όποιον θέλει. Ε, Έπρεπε να το είχα αναφέρει νωρίτερα βέβαια. Εγώ που γενικά δεν πίνω αλκοολούχα, απόψε θα μπορούσα. Πήγαινα να πω, είναι η τελευταία φορά που σας βλέπουμε, αλλά καλύτερα να μην το πω γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ μιλες ποτέ και τέτοια. Εκτός και αν ξέρετε εσείς κάτι, λέει ο κύριος Κίνγκ. Όχι, με χαρά λοιπόν σας βλέπουμε εδώ σήμερα. Πέμπτη συνεδρίαση διαλόγου ασφαλείας ή μη τι άλλο η τελευταία πριν τι εκλογέ για τον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα γίνει αξιολόγηση για την ε, Ένωση Ασφάλειας. Αυτά έχω να πω εγώ εισαγωγικά. Χαίρομαι που έχουμε εδώ τον ε, Julian King. Θα μας ενημερώσει, θα γίνει μετά η συζήτηση και η δεξίωση. Καλά κάνω και τα λέω ότι έχουμε ένα πιόμα. Ξέρω ότι δεν δείχνετε πολύ ενθουσιασμό. Σας παρακαλώ. Εσύ σε παρακαλώ, Λίβια. Έχει ξετρελαθεί, θα έρθει. Ωραία, ωραία, ωραία. Άντε λοιπόν να επιταχύνουμε, λέει ο κύριο Κίνγκ. Να επιταχύνουμε. Ήταν δύσκολη μέρα σήμερα. Εγώ τουλάχιστον ταλαιπωρήθηκα. Δεν τα, δεν τα μάθατε? Καλά, δεν θα σας τα πω. Με χαρά. Καλωσορίζω λοιπόν τον Επίτροπο για τα θέματα της ασφάλειας. Ε, πολλά θέματα έχετε. Τζούλιαν, αλλά πάρεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Άκουσα, διάβασα πριν ότι κάποιο ανακοινωθέν έλεγε πέμπτη και τελευταία ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο των Ορμόδιων κτλ. Ας πούμε τελευταία προγραμματισμένη, αν δεν έχετε αντίρρηση. Και πάντως ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή τη συζήτηση μαζί σα σήμερα. Την πρόσκλησή σα. Θα κάνουμε μια, έναν απολογισμό της προόδου της Ένωσης για την Ασφάλεια. Και εσείς το είπατε. Λίγος χρόνος μας μένει μέχρι ότου έρθει το, πέρος, το πέρας της τρέχουσας βουλευτικής περίοδου και άρα έχουμε να κλείσουμε ορισμένα θέματα, θα τα συζητήσουμε αυτά, σας πω τι έχουμε κάνει ακόμα, ήδη, τι ακόμα μένει να γίνει. Αν ε, με αντέξετε θα σας πω και μερικά ε, που βλέπω στο μέλλον ως προκλήσεις που πρέπει να μας απασχολήσουν. προκλήσεις για μια αποτελεσματική γνήσια ένωση ασφάλειας. Τι έχουμε επιτύχει λοιπόν καταρχάς. Και τι μένει ακόμα να γίνει, βράχει πρόθεσμα, τι πρέπει να μας απασχολήσει πιο συγκεκριμένα στο απότερο μέλλον. Ξεκινώ όμως λέγοντας ένα ευχαριστώ. Ευχαριστώ διότι με τη δική σας τη συνδρομή μπορέσαμε να κάνουμε πολλά. Και μάλιστα πρόσφατα πολλά. μπορέσαμε στο θέμα που αφορά το χώρο μας στον οποίο δραστηριοποιούνται οι τρομοκράτες να καταλήξουμε σε συμφωνία για τη διαλειτουργικότητα που ψηφίσατε εσείς νωρίτερα σήμερα. Πολύ σημαντικές αποφάσεις. Έτσι τα συστήματα ανταλλαγή πληροφοριών θα είναι πολύ πιο καλά, θα συνεργάζονται καλύτερα, πάντα με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. τα υφιστάμενα συστήματα ε, αλλά και τα νέα, τα αίτια στα έκρη, στη φυσέξιτ, θα διαφυλαχτούν αλλά θα μπορούν πια να συνομιλούν το ένα με το άλλο ή τα, όλα μεταξύ τους και πιο αποτελεσματικά έτσι ώστε οι πολύτιμες πληροφορίες που ήδη έχουν ε, εισαχθεί στα συστήματα αυτά να μην περάσουν απαρατήρητες, να μην μείνουν αναξιοποιητές. Και έτσι θα μπορούν οι αρμόδιοι να κάνουν τη δουλειά τους αξιοποιώντας τα και να προστατεύουν την ασφαλεία μας. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τη συνδρομή σας στα θέματα αυτά, τους συνεισηγητές Λέναρς, Μέλλερ. Εξαιρετική δουλειά, εξαιρετική συνεργασία μέσα σας. Και συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε και τους κανόνες για τις ε, πρόδρομες ουσίες που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες για να φτιάξουν ε, βόμβες με τις φωνικές τους συνέπειες στις χώρες στις πόλεις μας. Ευχαριστώ τον κύριο Μίκινς για την εξαιρετική δουλειά. Επίσης, ε, συμφωνία είχαμε για την πρόσβαση στις, στις χρηματοπιστωτικές πληροφορίες, πάλι πολύ σημαντικό να πλήξουμε το πορτοφόλι του τρομοκράτη, τον τρόπο με τον οποίο οργανώνει, δικτυώνεται, προβλέπει την τρομοκρατική επίθεση. Δύσκολες συζητήσεις, αλλά τα καταφέραμε. Και επίσης, προσωρινή συμφωνία είχαμε σήμερα για τη, για τη διαφύλαξη των στοιχείων ασφαλείας των ε, δελτίων ταυτότητας και την αποτροπή πλαστογράφησης ή υποκλοπής ταυτότητας για να μην μπορούν να κυκλοφορούν με πλαστές ταυτότητες οι τρομοκράτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα γίνει πιο ασφαλής λοιπόν η Ένωση έτσι και ταυτόχρονα οι πολίτες θα διατηρήσουν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας με αξιόπιστα έγγραφα ταυτότητας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα στον κύριο Πρέσβο από τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε. Σε προηγούμενα επεισόδια, όπως λένε σε αμερικανικές σειρές, είχαμε θέματα σχετικά με τα πυρομαχικά, με τη δυνατότητα κυκλοφορίας των τρομοκρατών, με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, με την ενίσχυση του δικτύου, του πλαισίου μάλλον για την αγορά, των έλεγχο των πυροβόλων, την ομοποίηση παρανομών εσόδων, την οδηγία PNR για τα στοιχεία επιβατών, αεροπορικών πτής, αεροπορικών ενέργειας κυκλοφορίας. Όλα αυτά λοιπόν έχουν προχωρήσει και ευχαριστώ όλους τους ε, βουλευτές που συνεργάστηκαν σε αυτά. Κυβέρνο έγκλημα. Συμφωνία σε συνεργασία με πολλές επιτροπές εξασφάλιστηκε ως προς το νομοθέτημα για την κυβερνό ασφάλεια. Συνιστατά αυτή τη στιγμή υπηρεσία κυβερνοασφάλειας, με συστήματα πιστοποίησης για την ενίσχυση του επίπεδου της κυβερνοασφάλειας, για τις διαγραμμικέ διαγραμμικές υπηρεσίες και την αντιμετώπιση μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπισοδίων. Συμφωνία είχαμε επίσης σε σχέση με νέους κανόνες για την κατά της απάτης και των ε, πατηλών πληρωμών σε μετρητά, ασφάλεια δικτύων ε, με την οδηγία νης, θεμέλιο λίθο της μελλοντική μας κυβερνοασφάλειας, μέτρα για την καλύτερη αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, πιέσαμε και τις ε, πλατφόρμες του διαδικτύου για ε, βελτίωση της αξιοπιστίας τους και των αλγορίθμων τους. Αυτά λοιπόν θα τα ξαναδούμε. Να φέρουν καρπούς και ενώπιση των ευρωεκλογών. Και βεβαίως ακόμα περισσότερα μένουν να γίνουν, όπως είπαμε, ιδιαίτερα στις ε, αμέσως προσεχείς εβδομάδες. Έχουμε μια πρόταση για κανονισμό για το παράνομο τρομοκρατικό περιεχόμενο που διατίθεται στο διαδίκτυο είναι ακόμη ένας, ε, ένας τομέας προτεραιότητας. Σας το έχω ξαναπεί άλλωστε, πρόκειται για περιεχόμενο το οποίο αποτελεί πραγματική απειλή. Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια είδαμε ότι κάθε τρομοκρατική επίθεση που έγινε στην Ευρώπη είχε και δομή μέσα από το διαδίκτυο και για, τη συνεργασία και για, για το συντονισμό αλλά και για την προβολή των τρομοκρατικών υποθέσεων, ε, επιθέσεων και βέβαια έτσι δηλητηριάζονται οι νέοι μας με το μικρόβιο της τρομοκρατίας. Ε, είπαμε ότι υπάρχει μια πλατφόρμα με συνεργασία εθελοντικής βάσης, ωστόσο πολλά ακόμα μένουν να γίνουν και μπορούμε να καταλήξουμε, ελπίζουμε, ε, σε μια συμφωνία σε κανονισμό προτινόμενο για να πατάξουμε με σαφείς κανόνες αλλά και διασφαλιστικές δικλείδες την κυκλοφορία αυτού του παράνομου τρομοκρατικού περιεχομένου. Ηλεκτρονικά στοιχεία, πιστήρια, αποδείξεις για την καταπολέμηση πάντα της τρομοκρατίας και της σοβαρή εγκληματικότητας. Είναι ένα θέμα που έχουμε σε εκκρεμότητα. Περαιτέρω προσπάθειες χρειάζονται ως προς το σύστημα ενημέρωσης ε, θεωριστιβατηρίων ε, με καλύτερη έρευνα του ιστορικού των ετουμένων θεώρηση, τεχνολογία, κυβερνοασφάλεια με το σχετικό κέντρο το ευρωπαϊκό αλλά και τα εθνικά κέντρα συντονισμού, πιστοποίηση δηλαδή, πρότυπα κτλ. Και πρέπει να συνεχιστεί και η δουλειά που κάνουμε για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, κυρίως εν ώψη των ευρωεκλογών του Μαΐου δουλειά που πρέπει να κάνουμε όλοι από κοινού. Εμπλέκονται πολλοί παράγοντες, πολιτικά κόμματα, υποψήφοι, κρατή, μέλη, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, οι πλατφόρμες του διαδικτύου. Πρέπει όλοι να συνεργαστούμε για να εξασφαλίσουμε πρόοδο και ιδιαίτερα οι πλατφόρμες πρέπει να προχωρήσουν περισσότερο και ταχύτερα ως προς την υλοποίηση του κώδικα συμπεριφοράς, καλή συμπεριφοράς για την από διάρθρωση αυτής της ε, προσπάθειας παραπληροφόρησης μέσα στο διαδίκτυο. Κάναμε και ένα εργαστήριο που συνομιλήσαμε εδώ στο Κοινοβούλιο απόψε για τα θέματα αυτά. Την Πέμπτη έχουμε ακόμη και εσείς νομίζω έχετε συμβάλει, Κλοντ, στην οργάνωσή του. Ένα άλλο εργαστήριο που θα περιγράψουμε την πρόοδο που χρειαζόμαστε για τα θέματα αυτά. Ωστόσο δεν μπορούμε να σταματήσουμε την πορεία μας, δεν μπορούμε να σταματήσουμε στο χρονικό σημείο των ευρωεκλογών, γιατί πρέπει να κοιτάξουμε και τις μελλοντικέ ανάγκες σε όρους ασφάλειας και μετά τις ευρωεκλογέ, νέα ζητήματα που θα προκύψουν με το νέο Κοινοβούλιο και τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και άρα πρέπει και να συνεχιστούν οι ε, συνομιλίες για τις μελλοντικέ πτυχές του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Πράγμα το οποίο σημαίνει επίσης και εδώ πολύ προσοχή έχουμε δώσει τελευταίες εβδομάδες στο θα βελτιωθεί η προστασία των ψηφιακών υποδομών. Ασφάλεια δηλαδή των κρατικών μηχανισμών, των επιχειρήσεων, της βιομηχανικής έρευνας, πνευματικής οκτησίας, επιχειρηματικών ε, ε, μοντέλων και σχεδίων, αλλά και δημοκρατικών θεσμών αλλά και προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Γιατί αυτό σημαίνει ταυτόχρονα προστασία την ε, βασική διάρθρωση της ζωής μας στη σύγχρονη εποχή. Όχι μόνο το 5G που μας απασχολεί τόσο το τελευταίο καιρό, αλλά και το νέφος, τα συνδεδεμένα ε, μηχανήματα, τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε, πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να συνεχίσουμε στην Ευρώπη όπως γίνεται τώρα να βλέπουμε να χάνονται οι τεχνολογίες εχμής από την Ευρώπη. Αν θέλουμε να επιτρέψουμε να αναπτυχθεί το φάσμα 5G χωριστά από τα κράτη-μέλη και τις επιχειρήσεις τους χωρίς συντονισμό, ή αν πρέπει να βρούμε κάποιες καλύτερες λύσεις. Ένα καλύτερο συντονισμό που θα βοηθήσει και στις ε, συλλογικές μας επενδύσεις με τέχνητη νοημοσύνη, το υπολογιστικό νέφος, τη ρομποτική κτλ. Όλα αυτά λοιπόν είναι περίπλοκα θέματα που σημαίνουν και αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο. Δεν θα είναι εύκολες οι λύσεις που θα δοθούν, αλλά πάντως έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Πρέπει να κοιτάξουμε το ψηφιακό οικοσύστημά μας, τη μεγαλύτερη διαφάνεια που πρέπει να εξασφαλίσουμε για να δούμε αν υπάρχει τρόπος να περιορίσουμε τους κινδύνους για την ασφάλεια με ένα δίκτυο ή αν απλώς υπάρχουν κίνδυνοι, υπάρχει μάλλον, έχει τέτοια σημασία μια συγκεκριμένη τεχνολογία που θα αποτελεί τη βασική δομή που δεν μπορούμε να τη θέσουμε σε κίνδυνο και άρα οι επενδύσεις πρέπει να περιοριστούν στην Ευρώπη και επίσης πρέπει να δούμε πόσο οι οικονομίες και η καθημερινή μας ζωή θα διαρθρωθεί πάνω σε αυτή την ψηφιακή οικονομία. Πολύ δουλειά τους επόμενους μήνες και τα χρόνια. Δεν θα είμαι εγώ αρμόδιος επαόριστον, αλλά όσο έχω αυτά τα καθήκοντα, μπορείτε να, στηρίζετε, να στηρίζεστε πάνω μου για τη συζήτηση, για τη συνεργασία. Είμαι απολύτως πεπισμένος ότι η Επιτροπή σας είναι το κατάλληλο όργανο και ε, έχει την ε, εμπειρία, την, ε, την ισορροπημένη προσέγγιση, τις ικανότητες να προωθήσει όλα αυτά τα θέματα. Το έχω δει στη συνεργασία μου μαζί σας έχετε μια πολύ διεξοδική, συνολική, ισορροπημένη προσέγγιση για όλα τα ζητήματα. Με τη συνεργασία του τα θεσμικά όργανα έχουν εξασφαλίσει σημαντική πρόοδο και ας μένουν αρκετά ακόμα πρέπει να ε, επιτευχθούν για να κατασκευάσουμε αυτή την ε, Ένωση Ασφάλειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολλά θέματα θίξατε, ενώ στο Συμβούλιο εσωτερικών ε, την προηγούμενη εβδομάδα. Το μόνο που συζητήθηκε ήταν πότε θα εφαρμοστούν ε, τα σχετικά συστήματα. Ε, πάντως ήταν πολύ καλό που αναφερθήκατε στο τι κάνει το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραίος ο κατάλογος που μας δώσατε. Συμμετρικός. Εκείνοι ακόμη μας ρωτούν για το PNR, ε, ενώ και εμείς ε, τους ε, ρωτάμε τα ίδια πράγματα. Έχουμε ένωση για την ασφάλεια και όλοι ασχολούνται με τις διάφορες πτυχές συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αναφερθήκατε και σε κάποιους από τους τριμερείς ε, διαλόγους και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ για όλη τη δουλειά σας. Ε, δεν θα ήθελα να ακούγομαι σαν να ε, έχουμε φτάσει στο τέλος του κόσμου. Τίποτα δεν είναι οριστικό στο κάτω-κάτω. Άλλωστε, ολονών μας η θητεία λύγει τώρα. Σας ευχαριστώ πάντως, διότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η επισκόπηση που μας δώσατε. πολύ συναρπαστικά τα στοιχεία που μα δώσατε. Ίσως συναρπαστικά να μην είναι και η κατάλληλη λέξη, ενδιαφέροντα τέλο πάντων. Μα γιατί με κοιτάτε έτσι. Ε, ναι, έχουμε πολλά θέματα τελευταία στιγμή. Έχουμε τη διαλειτουργικότητα, τι ε, προδρομέ ουσίε για κριτικές ύλε ε, κλπ. Υπάρχουν παρατηρήσει. Ε, παρακαλώ, κυρία Στίβεν Χέλγα και μετά ο κύριο Φρανς. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Κίνγκ, σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ για άλλη μια φορά. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για όλη την εξαιρετική δουλειά που έχετε κάνει. Γνωρίζετε ότι ήμουν συνεισηγήτρια στην ε, Επιτροπή ΤΕΡ και το 2018 Όσον αφορά την απορριζοσπαστικοποίηση, αναφέρθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε κατάλογο των δράσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε υπάρχουν σχετικοί δείκτες σχετικά με το πόσο επιτυχή είναι τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται. Ζητήσαμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει τι γίνεται με τους πόρους αυτούς ε, που ε, διατίθενται για την απορριζοσπαστικοποίηση. Τι ποσά δηλαδή έχουν δοθεί στα διάφορα προγράμματα. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι... Όσον αφορά μια αρχή για την απορριζοσπαστικοποίηση, τι συγκεκριμένη χρηματοδοτική ή πρακτική υποστήριξη μπορεί να παρεσχεθεί. Σας ευχαριστώ. Λίβια Ρόκα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη δουλειά που έχετε κάνει. Έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά και στον τομέα της ασφάλειας. Πολύ χρήσιμη η δουλειά που έχετε κάνει πάνω σε αυτό το δύσκολο έγγραφο. Όσον αφορά δε την κυβερνοασφάλεια, γιατί σε αυτήν αναφέρομαι, καθώς και τις ψηφίσει ειδήσει, ε, τα fake news, πρόκειται για πολύ σημαντικά θέματα. Αναφερθήκατε στα πιο βασικά ζητήματα του χαρτοφυλακίου σας. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ σε ένα θέμα που αναφέρεται σήμερα στον τύπο. Πρόκειται για μια εκστρατεία της Ουγγαρίας, την οποία η Επιτροπή αποκαλεί ψευδείς ειδήσει, fake news. Εγώ δεν είδα τίποτα ψευδές. Θα ήθελα να ακούσω όμως και τη δική σας άποψη. Διότι μόλις έδωσα συνέντευξη και είναι πολύ δύσκολο θέμα, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να δαπενήσουμε άλλο χρόνο σε αυτό. Πρέπει να επικεντρωθούμε στα θέματα που αναφέρατε εσείς εδώ σήμερα προς όφελος ε, των πολιτών μας και για να ε, διασφαλίσουμε την ασφάλειά τους. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Φράνς. Αγαπητέ Τζούλιαν Κίνγκ και από πλευράς των Πρασίνων ε, θα ήθελα να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας ε, για τον τακτικό διάλογο και την καλή συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Ωστόσο, ακόμη αναρωτιόμαστε τι μέτρα έχουμε αναλάβει, πόση ασφάλεια έχουμε πετύχει και με τι κόστος, μήπως θα μπορούσαμε τους ε, διαθέσιμους πόρους να τους ε, χρησιμοποιήσουμε με άλλο τρόπο. Σήμερα το πρωί η Επιτροπή μας ψήφισε τη δέσμη μέτρων για τη διαλειτουργικότητα. Κάτι που ε, συνδέεται με πολλά μέτρα των τελευταίων ετών που έχουν ένα κοινό. Την συλλογή πολλών δεδομένων αθώων ανθρώπων, κάτι που στοιχίζει και πάρα πολύ. Αυτό καταρχάς είναι αντισυνταγματικό, όπως έχει αποφασίσει ήδη δύο φορές το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μία τρίτη φορά όσον αφορά τα δεδομένα επιβατών. Δεύτερον, ε, αυτό στοιχίζει δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία μας λείπουν σε άλλους τομείς. Και τρίτον, ε, δεν μας βοηθάει να βρούμε την σωστή λύση. Επίσης, ε, έχουμε τη διασυνοριακή δίωξη ε, σε περίπτωση κανονικών ε, εγκλημάτων, αλλά και σε περίπτωση οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατίας. Θα πρέπει να κινούμαστε στα πλαίσια του κράτους δικαίου. Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία ε, εάν επιτρέπουμε στις αρχές να ζητούν στοιχεία από την εταιρεία παροχής τηλεφωνίας μου στην ε, Γερμανία, αυτό είναι πρόβλημα όσον αφορά την ασφάλεια και όχι λύση, αν κοιτάξουμε και την κυβέρνηση στη Βουδαπέστη. Ασφάλεια σημαίνει κυρίως ασφάλεια, διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και της ελευθερίας με αυτό το πνεύμα σφίγουμε από την αίθουσα σήμερα. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο μέλλον, κύριε Επίτροπε. Η, Τερίδα, η Τερέσα Μπεθερίλ. Ευχαριστώ πολύ. όλες ε, τις παρεμβάσεις σας τις εκτίμησα, πάντοτε δείξατε διαθέσιμος ε, και με πολύ μεγάλη χαρά συνεργαστήκαμε μαζί σας. Είστε απόλυτα δεσμευμένος ε, και προσιλωμένος στα θέματα της ασφαλείας. Ε, δυστυχώς ενίοτε η μνήμη μας είναι πολύ βραχία και μόνο όταν γίνεται μια τρομοκρατική επίθεση όλοι μας βάζουμε τα διάφορα ε, πανό, κονκάρδες, είμαι, είμαστε όλοι Παρίσι, είμαστε όλοι Βρυξέλλες κτλ. κτλ. Αλλά ε, πρέπει να πω ότι και αυτό αρχίζει να ε, ξεχνιέται μετά από όχι 15 μέρες ίσως που γίνονται στην αρχή, αλλά και μετά από μια εβδομάδα. Ε, θα ήθελα να μιλήσω για την αντιτρομοκρατική στρατηγική και για την προστασία στα θύματα. Προστασία, πρόληψη, δίωξη των δραστών, των τρομοκρατών και ε, φροντίδα στα θύματα. Αυτές είναι τέσσερις λέξεις. Ε, δεν μπορώ να συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα, δυστυχώς, διότι είναι πολύ εύκολο να λέμε ότι πρέπει να προλάβουμε. Ε, και ότι πρέπει να προστατεύουμε τα θύματα και ότι πρέπει να αποφεύγουμε τις επιθέσεις. Ε, αλλά ταυτόχρονα είμαστε κατά του PNR, ε, της Συμφωνίας για τη Συλλογή Δεδομένων. Πράγματι μπορεί να μην χρησιμεύουν τα στοιχεία που συλλέγουμε τους περισσότερους και όμως χρησιμεύουν τελικά γιατί αν δεν έχουμε στοιχεία για τα ταξιδιωτικά δεδομένα, κάποιο που πηγαίνει ή έρχεται από τη τα κτλ. μπορεί να μην έχει κάνει το έγκλημα εν συγκεκριμένο συγκεκριμένο άτομο. Όταν το έχει κάνει όμω θα υπάρχουν ήδη θύματα. Πού είναι η πρόληψη, πού είναι η προστασία επομένω. Γι' αυτό θεωρώ ότι τα μέτρα είναι δίκαια. Η διαλειτουργικότητα ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό που η Επιτροπή Ειδική ε, για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας ε, το είχε ζητήσει ε, για όλες τις χώρες από τις οποίες μεταβήκαμε. Είναι πολύ καλό που έχουμε αυτή την οδηγία. Σίγουρα χρήζει βελτίωσης, όμως νομίζω ότι Αυτά τα έτη δυστυχώς ε, στιγματίστηκαν από τον Πατακλάν, ε, το Εσβρυξέλλε, τη Βαρκελόνη, το Λονδίνο ε, και τις τρομοκρατικές εκεί επιθέσεις. Ίσως ε, δεν ε, προλάβαμε, αλλά σίγουρα έχουμε σημειώσει πρόοδος ό,τι αφορά την ε, προστασία. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Κίνγκ γιατί είναι μεγάλη συμβολή του για την προστασία ακριβώς στα θύματα και την πρόληψη τέτοιων επιθέσεων. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ο Πρόεδρος, θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Αν μου επιτρέπετε, να θέσω ένα φιλοσοφικό ερώτημα. 5 και 33 το απόγευμα την Τετάρτη. Τετάρτη? Α, όχι, Τρίτη. Τι έχω πάθει και ξεχνάω. Τέλος πάντων, λοιπόν. Τι διδάγματα θα αντλούσατε. Έχουμε τον διάλογο για την ασφάλεια. Τον τελευταίο πριν τη λήξη της θητείας από ό,τι φαίνεται. Είστε ο πρώτος ε, αρμόδιος για θέματα ασφάλειας επίτροπος και συνεργάζεστε με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που βέβαια ε, έχει στο παιδί δηλαδή, τον σε ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων και μεταξύ άλλων προστασία δεδομένων που είναι ευρύ πεδίο. δεδομένων των συστάσεων του Συμβουλίου, δεδομένων του γεγονότος ότι πρόκειται και θα είναι εθνική αρμοδιότητα οι υπηρεσίε τα κτλ. Υπάρχουν κάποια διδάγματα ευρύτερα. Είναι ευρύ το ερώτημα και όπως το θέτω και λοιπόν λυπάμαι που σας ρωτώ, αλλά είστε ο πρώτος εσείς ε, Επιτρόπος για θέματα ασφάλειας. Υπήρχαν συγκεκριμένα ζητήματα και άρα εστιάσαμε σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα εδώ, αλλά υπάρχει και το θέμα των θεμελιών δικαιωμάτων, της των δεδομένων, που είναι ευρύτερα ζητήματα, όπως και η διασυνοριακή ευθύνη και αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα επίμαχο πάντοτε ζήτημα. Ίσως όχι τόσο επίμαχο εμφυλεγόμενο, αλλά σίγουρα συζητήσιμο. Ως Επίτροπος λοιπόν αρμόδιος για θέματα ασφαλείας, ε, τι δίδαγμα έχετε ε, αντλήσει. Ίσως ότι καλό είναι να υπάρχουν κάποιοι φάκελοι συγκεκριμένοι για να τους επικραστούμε, δεν ξέρω. Σα ε, απαντήσετε παρακαλώ. Ο κύριος Κίνγκ, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους βουλευτές που συνεχίζουν να ασχολούνται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό εάν ε, θέλουμε να προασπίσουμε τις ευρωπαϊκές μας αξίες. Γιατί για να το κάνουμε αυτό πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε και ικανοί να προστατεύσουμε τους πολίτες και να διαχειριστούμε ορισμένους από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν. Για την κυρία Στίβενς ε, που μίλησε για την Επιτροπή ΤΕΡ και το έργο της, δηλαδή, δηλαδή Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας. Ε, θα απαντήσω και στον πρόεδρο τη Επιτροπή Λίμπε, γιατί είμαστε στην Επιτροπή Λίμπε. Θέλω όμω να σα ευχαριστήσω και εσά προσωπικά, κυρία Στίβενη, και όλου όσοι συμμετείχαν στο έργο τη Επιτροπή ΤΕΡ και ε, για την έκθεση που συνέταξε. Είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό κείμενο. Σίγουρα αντλεί σωστά διδάγματα και προτείνει μέτρα και τρόπους ε, προς τα εμπρός για την αντιμετώπιση της ε, τρομοκρατίας και την ε, πρόληψη και ελπίζω την φροντίδα στα θύματα, την προστασία των θυμάτων. Στο, στην αρχή του έργου σας θα περίμενε κανείς ε, να μην είναι και τόσο ε, θετικό απέναντι στα πέρασμα της έκθεσης στην άτυπη συνεδρίαση τα κράτη-μέλη όμως αναγνώρισαν τη σοβαρότητα του έργου της Επιτροπής ΤΕΡ, αναγνώρισαν τη σημασία των συμπερασμάτων σας και των συστάσεων που διατυπώνετε για το μέλλον. Ο διάλογος μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων, το Κοινοβούλιο είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ενίοτε ε, μπορεί να είναι και πολύπλοκος αυτός ο διάλογος όπως το γνωρίζετε. Πάντως σας πιστώνετε, πιστεύω το γεγονός ότι σε αυτό τον επίμαχο τομέα τελικά πήρε ε, θετική υποστήριξη από το Συμβούλιο η εκθεσή σας και οι συστάσεις σας, ό,τι αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ρίζος παστικοποίησης. Πάρα πολύ σωστά είπατε ότι αν θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο στο μέτωπο αυτό, θα πρέπει να έχουμε μια επισκόπηση κατάστασης και να θέσουμε ε, στους εαυτούς μας τα σωστά ερωτήματα. Μετά από κάποια σχόλια και από το Κοινοβούλιο αλλά και από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αποφασίσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως θα πρέπει να δημοσιοποιήσουμε τις εσωτερικές αυτές ε, επισκοπήσεις ε, της πολιτικής μας. Εγώ θα προτιμούσα να είχε γίνει αυτό λίγο νωρίτερα, αλλά καλύτερα αργά παρά ποτέ και όταν θα είναι δημοσιοσία διαθέσιμα αυτά τα έγγραφα, ίσως θα έχετε στον διαδοχό μου να θέσετε κάποιες ερωτήσεις και για το πόσο αποτελεσματικά είναι αυτά τα μέτρα. Για να απαντήσω στην ερώτησή σα για την πρόοδο. Εγώ νομίζω ότι έχουμε επιτύχει πρόοδο και είμαι υπερήφανο για τη στήριξη που συνεχίζουμε να παρέχουμε στι ε, χώρε και στους φορεί που είναι στην πρώτη γραμμή που καθημερινώς αντιμετωπίζουν το, την πρόκληση της ριζοσπαστικοποίησης ε, με το ΡΑΝ και άλλα δίκτυα. Όμως, κάτι ακόμη που έχει γίνει τώρα είναι ότι αυτή η εμπειρία ε, στη βάση, στην πρώτη γραμμή, έχει συντονιστεί καλύτερα με τις τοπικές διοικήσεις, ε, τους εθνικούς αρμόδιους φορείς. Και αυτό είναι κάτι ευπρόσδεκτο, γιατί αν θέλουμε να έχουμε μια αποτελεσματική πολιτική, αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί με από τη βάση, αλλά να έχει και την δέουσα πολιτική υποστήριξη. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θετικό βήμα το οποίο έχουμε κάνει. Σε ό,τι αφορά τις ψευδείς ειδήσει. Αυτό το τελευταίο που είπατε δεν το ε, έχω υπόψη, έχω διαβάσει όμως κάποιες ε, αναφορές παλαιότερες. Οι ψευδείς ειδήσει ότι χρησιμοποιούνται ως ένας πολιτικός όρος ε, για τη διατύπωση σχολείων για διάφορα ε, απόψεις, συνήθω από τον οποίο δεν συμφωνεί κάποιος, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το έργο που έχει γίνει. Από την περσινή άνοιξη για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων και για να ορίσουμε την παραπληροφόρηση. Γιατί πρέπει να αποφύγουμε να μπούμε σε μια ευρύτερη συζήτηση με την οποία μπορεί κανείς να συμφωνεί ή να μην συμφωνεί. Παραπληροφόρηση που έχουμε ένα πολύ σαφή συγκεκριμένο ορισμό που είναι εσκεμμένη διάδοση ψευδών πληροφοριών για οικονομικό ή πολιτικό όφελος. Θέλουμε λοιπόν να προωθήσουμε ορισμένα μέτρα με το Κοινοβούλιο, με τους υποψηφίους, με τα κράτη-μέλη και τις πλατφόρμες των κοινωνικών μέσων, ε, με στόχο ακριβώς την παραπληροφόρηση, είναι ζωτική σημασία στο έργο αυτό, ιδίως ε, εν ώψη και των ευρωεκλογών και θα συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά που κάποιες φορές βέβαια που μας οδηγεί σε ένα είδος πολιτικής συζήτησης με τους διαφωνούντες. Ανθρώπους έχουν διαφορετικές απόψεις. Εγώ όμως θέλω να εστιάσουμε συγκεκριμένα στα μέτρα που πρέπει να λάβουμε για να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση όπως την έχουμε ορίσει. Για το ερώτημα του κύριου Φραντς για την δέουσα χρήση την ορθή χρήση των μέσων και εργαλείων. Είτε είναι η βάση δεδομένων, είναι το ΣΥΣ, το σύστημα πληροφοριών, οτιδήποτε άλλο έχουμε συμπεριλάβει στο πλαίσιο της εργασίας μας για την ασφάλεια. Εγώ συμφωνώ μαζί σας πως πρέπει να φροντίσουμε τα μέσα και εργαλεία, τα μέτρα που λαμβάνουμε, ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά για τους στόχους για τους οποίους έχουν δημιουργηθεί. Αν κάποιος, μια διοίκηση ή οποιοδήποτε προσπαθεί να χρησιμοποιήσει με εσφαλμένο τρόπο καταχρηστικά ε, τα μέσα αυτά για άλλους σκοπούς από αυτούς για τους οποίους νομίμως προορίζονται. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ξεσκεπάσουμε και να ασκήσουμε κριτική για την κακή χρήση, για την κατάχρηση αυτών των μέσων και εργαλείων. Δεν αρκεί δηλαδή απλά να ε, ελέγχουμε ότι χρησιμοποιούνται σωστά αυτά τα μέσα και εργαλεία. Σε ό,τι διαφορά την απόπειρα κατάχρηση αυτών των μέσων, του ΣΥΣ για παράδειγμα, ήταν ελάχιστε οι φορές και όταν έγινε υπήρξε κατακραυγή. Και αυτό το θεωρώ θετικό. Διότι δείχνει ότι αυτά τα εργαλεία είναι κατανοητά και ο κόσμο θέλει τα χρήματα που έχουν δοθεί προ αυτό το σκοπό να χρησιμοποιούνται σωστά και για το σκοπό αυτό και όχι να υπάρχει κατάχρηση. Για την κυρία Μπεθερίλ, είπατε δύο πράγματα πολύ σημαντικά νομίζω. Το πρώτο είναι ότι πρέπει ε, να διδαχθούμε ε, από την πολιτική που ε, έχουμε εφαρμόσει μέχρι τώρα, αλλά όχι πράγματι να σπέβδουμε, να δράσουμε αμέσως μετά από μια φρικτή επίθεση ε, και μετά να ξεχαστούμε και να τα παρατήσουμε όλα. Αν θέλουμε να γίνει πρόοδος, ε, θέλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω στα θέματα, ακόμα και αν δεν είναι πλέον πρώτο σέλιδο η πρώτη είδηση στην τηλεόραση. Έτσι θα μειώσουμε και το... τις πιθανότητες να ξαναμπούν σε κάποιο πρωτοσέλιδο αντίστοιχες, ε, αντίστοιχες ειδήσει σίγουρα πρέπει να διατηρηθεί η όθηση αυτή και να μην έχουμε ε, αυτά τα τους δύο χρόνους, αντίδραση σε δύο χρόνους. Γρήγορη δράση, μετά σταματάμε και ξεκινάμε αν ξανασυμβεί κάτι. Έχουμε την οδηγία για την αντιμετώπιση τρομοκρατία, με τι διατάξει για την φροντίδα στα θύματα. Με τη δική σα ενθάρρυνση, η Κομισιόν θέλει να δημιουργήσει και ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνη ε, για τα θύματα τρομοκρατία, φέτο κιόλα. Και ελπίζω αυτό να είναι αφετηρία για κάτι μεγαλύτερο. Και γνωρίζω πω ε, θα συνεχίσετε να μα ενθαρρύνετε προ αυτή την κατεύθυνση και προσβλέπω στην 11η Μαρτίου για να δείξουμε εκ νέου το σεβασμό μας στα θύματα των διαφόρων επιθέσεων, αντιλώντας και τα απαραίτητα διδάγματα για το μέλλον. Και επειδή μιλάμε για διδάγματα, για το μέλλον, ο Κλοντ με παρακάλεσε να πω κάτι ε, ως κατακλίδα των ε, εργασιών τα τελευταία αυτά χρόνια. Νομίζω ότι το είπα εξ αρχής και επαναεπιβεβαιώνεται αυτό από την εμπειρία μου. Μια αποτελεσματική πολιτική ασφαλής μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν είναι βαθιά ριζωμένη στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πρέπει η πολιτική να τα σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, η εφαρμογή και η επιβολή των μέτρων πρέπει και να σέβεται και να φαίνεται ότι σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλό ε, που ένας φορέας όπως ε, το eBay παίρνει μια προσέγγιση ε, συνεκτική απέναντι στα θέματα αυτά και έχετε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και ελπίζω να συνεχίσετε να τα βλέπετε από ένα ευρύτερο πρίσμα τα πράγματα. Είναι καλό αυτό για τη χάραξη πολιτική στον τομέα τη ασφάλεια. Θα σα να επίση να αποφύγετε αχρίαστε συζητήσει περί επικουρικότητα. Ποιο κάνει τι γιατί νομίζω ότι καταφέραμε κάπως να ξεπεράσουμε αυτή τη συζήτηση. Θα πρέπει να μιλάμε για αποτελεσματική χάραξη πολιτικής και αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικής. Θα υπάρξουν ζητήματα που θα είναι πολύπλοκα. Υπάρχουν ήδη πολύπλοκα ζητήματα, αλλά νομίζω ότι οι αρχές των κρατών μελών σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν δεχθεί ότι ναι, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Συχνά όμως η συνεργασία μπορεί να φέρει καλύτερο αποτέλεσμα, ιδίως σε ευρωπαϊκό δηλαδή επίπεδο παροχή υποστήριξη στα κράτη αυτά για να φέρουν σε πέρα στις διάφορες αρμοδιότητες και εκεί πρέπει να εμείνουμε στη συνεργασία και κατά το δυνατό να αποφύγουμε να τσακωνόμαστε για το ποιο κάνει τι. του λεχθέντος φυσικά και έχουμε ευθύνη και θα συνεχίσουμε να ε, ασκούμε υπεύθυνα το ρόλο μας. Είναι άλλωστε πράγματα που είναι δεσμευτικά για εμά και πρέπει να τα κάνουμε, άλλα είναι δεσμευτικά για τα κράτη-μέλη πρέπει να τα κάνουν. Το ίδιο ισχύει για του εκτελεστικού οργανισμού και πρέπει να έχουν βέβαια και την απαιτούμενη χρηματοδότηση για να μπορούν να φέρουν σε πέρα στα καθήκοντά του. Άρα η δική σα εστίαση στην υλοποίηση, στην εφαρμογή είναι κάτι πολύ θετικό και σημαντικό. Κάτι που ίσως θα μπορούσατε να το σκεφτείτε και για τη μελλοντική θητεία, για την επόμενη θητεία, είναι ο βαθμός φιλοδοξίας που θέλετε να έχετε για τη δημιουργία μιας ένωσης ασφάλειας. Κάναμε πολλή δουλειά, κάνατε εσείς ήδη πολύ πριν έρθω εγώ, αλλά και τα δύο τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την αντιμετώπιση των κλασικών κυβερνοαπειλών έχουμε κάνει πολλά. Και πρόσφατα για την κατάχρηση πληροφοριών που μεταδίδονται στον κυβερνοχώρο και την εσκεμμένη παραπληροφόρηση. Έχουμε κάνει πολλά, επαναλαμβάνω, και θα συνεχίσουμε. Όπως και για την αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Αν όμως δούμε το μέλλον, κοιτάξουμε προς τα εμπρός, υπάρχουν κάποιες προκλήσεις που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο, ιδίω, οι οποίες θα είναι πάρα πολύ σημαντικές για την εξασφάλιση της ασφάλειας. Και όπως κάνει το Συμβούλιο, όπως κάνει η Κομισιό, θα πρέπει και εσείς να δείτε πώς θα ενώσουμε τις κουκίδες σε ε, όλα αυτά τα θέματα που είναι συγκινούντα δοχεία κατά κάποιο τρόπο. Αν δεν τα δούμε έτσι θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες. Και αν δεν βρούμε μια κοινή προσέγγιση. Στο Συμβούλιο υπάρχουν ε, πολύ σοβαρά ζητήματα κυβερνοασφάλειας τα οποία συζητούνται στο Συμβούλιο Τηλεπικοινωνών. Όχι ότι έχω κάτι ε, ενάντια στο Συμβουλίο Τηλεπικοινωνιών. Αλλά υπάρχουν πολλά άλλα, πολλέ άλλε παράμετροι που την αληθούν υπόψη. Το Κοινοβούλιο ε, και χαίρομαι που έχω πάει σε διάφορες επιτροπές, αλλά έχω έρθει σε τρεις-τέσσερις επιτροπές που συζητούν ε, διαφορετικές πτυχές ε, της ψηφιακής ασφάλειας και της κυβερνοασφάλειας. Σας παρακαλώ λοιπόν αυτό να το σκεφτείτε, δηλαδή να δείτε πώς θέλετε να οργανώσετε τη συζητή σας στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και το κοινοβουλευτικό έργο. Για να δημιουργηθεί μια ένωση ασφάλεια σε έναν κόσμο όλο και πιο διασυνδεδεμένο και ψηφιακό. Δεν μπορώ να απαντήσω, είναι μια πρόκληση για τα κράτη-μέλη, για τα θεσμικά όργανα και για το κοινοβούλιο, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ. Και αύριο το πρωί έχουμε μια σχετική εκδήλωση. Θα συστήσουμε το hacking και άλλα θέματα τέτοια. Με την κυρία Σκοτ Κέιτο και τον Τζούλιαν Κίνγκ. Ομιλητές. Πολλή δουλειά που έχουμε να κάνουμε και ενώπιση των ευρωεκλογών βεβαίω που δεν εξαντλήσαμε σήμερα. Αλλά έχει αρχίσει η δουλειά, δεν έχει τελειώσει, αλλά έχει αρχίσει τουλάχιστον. Ευχαριστώ πολύ για όλη τη δουλειά με τους ε, εισηγητές μας, συνεργασία και τα λοιπά, το προσωπικό μας. Ιδιαίτερα στην Τζοάννα έχουμε δυναμία και εσάς σας συμπαθούμε πολύ βέβαια. Και έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά, όπως έλεγα, δύσκολα θέματα. Είπατε κι εσείς ότι οι συγκητές διαδέχονται ο ένας τον άλλον σε δουλειά. Και το προσωπικό μας νομίζω. Εξής συγχαρητηρίων. Είναι όμως, όπως είπαμε, λεπτά τα θέματα. η διαλειτουργικότητα του χερούν, πόσες ε, τροπολογίες δέχτηκες. Ούτε εσύ δεν θυμάσαι. Πολύ δουλειά λοιπόν. Ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστούμε όλους και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε με ένα ποτήρι που όμως προβλέπεται για τις 6.30 και ενημερώθηκα ότι μια και είναι εδώ κοινοβούλιο δεν μπορούμε να βγούμε και να το πιούμε πιο νωρίς το ποτό μας. Μόνο 6,5. Πρώτη φορά τελειώνει η συνεδρίαση με τη δική μου τουλάχιστον προεδρία πιο νωρίς. Άρα έχουμε να σκοτώσουμε χρόνο μέχρι τις 6,5 στο μπαρ του τρίτου εδώ στο ίδιο κτίριο που βρισκόμαστε. Δεν γίνεται να το πάμε λίγο πιο νωρίς. Καλά. Εγώ με τον Τζούλιαν πάντως θα πάμε εδώ στην πρασερή του, του τρίτου. Και όποιο θέλει ας έρθει. Δύο Βρετανοί στο μπαρ στις 6.30. Αν θέλετε, κουπιάστε. με τη βουλευτική μου αποζημίωση. Εγώ σας κερνάω. Ίσως και κάτι να τσιμπήσουμε. Ελάτε λοιπόν, κοπιάστε παρακαλώ. Και όπως είπα, αλκοόλ μπορεί να μην πίνω, αλλά θα χρειαστεί να πιω κάτι. Δύσκολη μέρα σήμερα. Σας ευχαριστούμε όλους. Και χαίρομαι ιδιαίτερος που έχουμε και τη διερμηνία εδώ και βλέπω τον ε, συνάδελφο το γαλλόφωνο να γελάει με τα αστεία μου με χρονοκαθυστέρηση. Όπως έλεγα, 6 και 30 στον Πράσερη. 30 λεπτάκια. Μιλάω όπως βλέπετε για να σκοτώσω το χρόνο. Έφαγα ακόμα τη 3 λεπτά. Άντε, μένουν άλλα 30 λεπτά για το ποτό. Ευχαριστούμε. Μέχρι τις 29 Μαρτίου μεσάνυχτα θα μας βρείτε στο μπαρ.